Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. You have been in favor, Mrs. Auta. Κυρία Χάουτα, είστε υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. Εκατόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Okay. have been, have been adopted? This has no, not been adopted? Not adopted. Not okay. My, my mistake, sorry, we are at 131. Λάθος μου, λάθος μου. Σε άλλη τροπολογία, στην 131 είμαστε υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 131. and that has been adopted. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Συμβιβαστική 1. Παναλαμβάνω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εναλλακτική συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω χέρια. Ψηφίζουμε την εναλλακτική συμβαστική 1. Απορρίπτεται. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 132. Εγκρίθηκε. 136 in favor. 136 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140. Περ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Adopted. 142. 142 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Okay, let's check on 11. Έλεγχος για την 11. Εγκρίνεται. Λόγω της κυρίας Χαουτάλα. Προσθέτουμε χειρονακτικά την κυρία Χάουταλα.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 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ δεύτερο τμήμα κατά αποχές απορρίπτονται 214. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 228 υπέρ κατά άλλη μια φορά παρακαλώ 228 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 230 υπέρ κατά άποχες έλεγχος για τη 230 παρακαλώ. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ κατά επανάληψη για τη 243 παρακαλώ υπέρ κατά Πρέπει να γίνει έλεγχος. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χαουτάλα υπερψηφίζει. Άρα εγκρίνεται. Μάλιστα. 244 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε τη 246 παρακαλώ. And that has been rejected. Απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σημαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 280 υπέρ 80 κατά. Τώρα είμαι σίγουρος πως ψήφισαν οι πράσινοι. Ξανά 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά επανάληψη παρακαλώ για την 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.94 υπέρ μαζί 2.94 2.98 και 300 υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται 306 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 307 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 38 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 38 παρακαλώ εγκρίνεται μαζί με την κυρία Χαουτάλα. 38 εγκρίνεται, 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ Συγγνώμη, έκανα λάθο, Ζεπρόδο. 324 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 336 υπέρ κατά 336 επαναλαμβάνουμε. 336 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά έλεγχος για τη 46 παρακαλούμε. απορρίπτεται. 337 και 338 υπέρ, κατά, έλεγχος για αυτές τις δύο. Απορρίπτονται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 346 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 347 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 ή 350 έως και 365 ψηφίζουμε από κοινού υπέρ τέσσερι σελίδε μονάχα στον κατάλληλο ψηφοφορία. Ξαναψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. λέει 60 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Αποχέ. αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ ζητώ συγγνώμη κύριε πρόεδρε. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α, α ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε για την 68. Ψηφίστε παρακαλώ. Απεριφθεί. Συμβιβαστική ΒΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ όχι λάθος ε, κατέπεσε 87 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφιστεί για την 87 παρακαλώ. That, Εγκρίνεται 87, 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Λάθος πάλι, κύριε ο Πρόεδρος. Έπρεπε να είχαμε πάει στην 111. Okay. 113. So... 113 για την ακρίβεια υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται, 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι λάθος, εγκρίνεται ε, η 120 εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 125 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε για την 125. Παρακαλώ but there Λάθος, λάθος, ε, ξεκάθαρα απερίφθη. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα για την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Και εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Τζαμπάνσκι, τον εισηγητή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε αποτελεσματικά. Είμαστε στο σημείο 13. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Διδιέ. Και παρακαλώ ησυχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με ιδιαίτερο ευτυχή που μπορώ να σα παρουσιάσω αυτό την προσχέδιο γνωμοδότηση. Δέκα μήνε μετά την ε, ένταξή μου μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω αναλάβει έναν φάκελο πολύ δύσκολο και σημαντικό και ευαίσθητο, το γνωρίζω και μάλιστα που έχει δημιουργήσει αντιθέσει. Με την ταπεινότητα που χρειάζεται ε, να προσεγγίσει κανεί ένα τέτοιο θύμα, δεν θα σα κρύψω ότι δεν ήταν πάντοτε εύκολο, γιατί υπήρχαν πολύ διστάμινε απόψει και σε ορισμένε περιπτώσει, θα έλεγα 100% αντίθετε μεταξύ του. Για παράδειγμα, όταν θα δεχτούμε να έχουμε συλλογικές προσφυγές ε, γενικού χαρακτήρα έτσι ώστε για παράδειγμα κάθε πολίτης ο οποίος ανέφτεψε ε, αέρα με ρήπους να αποζημιωθεί. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι το επιθυμούν 100% άλλοι οι οποίοι δεν το επιθυμούν. Όλοι αντιλαμβάνονται βέβαια ότι η λύση είναι η μέση οδός. Προσπάθησα να σεβαστώ τις ανησυχίες, ε, τις εύλογες που είχε ο καθένας και να προσπαθήσω και εγώ να βρω λοιπόν αυτή τη μέση οδό. Και αυτό σας παρουσιάζω σήμερα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσει που έχουν οι καταναλωτές και οι πολίτες και την προστασία των δικαιωμάτων ε, που τους οφείλουμε, αλλά επίσης για να προστατεύσουμε τις τίμιες εκείνες επιχειρήσεις που θα μπορεί να βρίσκονταν αντιμέτωπες με υπερβολικές ε, συλλογικές προσφυγές ε, κακή την πίστη, οι οποίε ε, ήταν στην πραγματικότητα εναντίον της ίδιας της έννοια των συλλογικών προσφύγων. Έτσι ώστε δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στου καταναλωτέ να έχουν πρόσβαση αποτελεσματική στη δικαιοσύνη χωρί να ακροτηριάσουμε την οικονομία μα. Με αυτή τη φιλοσοφία κινήθηκα και με αυτή τη φιλοσοφία προσπάθησα να, να συντάξω την γνωμοδίτησή μου όπως πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργούμε στο κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, οι συλλογικέ προσφυγέ θα πρέπει να μπορούν να ε, εφαρμόζονται όταν έχουμε παραβιάσει ε, που έχουν ευρείε επιπτώσει στου πολίτε μας. Έχουμε θέσει ένα λογικό όριο, δηλαδή να έχουν πληγεί 50 ή περισσότεροι πολίτες. Βέβαια αυτό μπορεί να τροποποιηθεί αυτό ο αριθμό. Ε, γιατί πιστεύω αν έχουμε μια προσφυγή η οποία στην πραγματικότητα αναφέρεται ή έχει πλήξει ή συντροπή, έχουν ένα συμφέρον μόνο λίγοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα δεν είναι συλλογική. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να εξετάσουμε μάλλον ποιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τέτοιε συνολογικέ προσφυγέ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι ενώσει καταναλωτών αναγνωρισμένε το οποίο σημαίνει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα επενδυτικά ταμεία ή τα δικηγορικά γραφεία, τα οποία θα μπορούσαν να καταχραστούν το, το σύστημα των συλλογικών προσφυγών και να καταντήσουμε σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη που διαπιστώνουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε, που δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που επιθυμούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια με τα οποία ε, περιγράφεται μια τέτοια ένωση και να συμπεριληφθεί σε αυτό για παράδειγμα το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση από τρίτους με την εξαίρεση βεβαίως των μελών τους. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε ενώσει καταναλωτών οι οποίε χρηματοδοτούνται από το κράτο με σημαντικέ επιδοτήσεις. Γνωρίζω βέβαια ότι αυτό δεν ισχύει σε άλλα κράτη-μέλη και ότι θα έλεγα ότι μάλλον είναι γαλλική εξαίρεση. Όμω τέτοια κριτήρια χρειάζονται επίσης νομίζω ότι χρειάζονται εχέγγυα για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης. Γιατί θα μπορούσαμε να φανταστούμε το ενδεχόμενο μια επιχείρηση συγκεκαλυμμένα να χρηματοδοτεί μια ένωση, έτσι ώστε εκείνη η ένωση με τη σειρά της να κάνει μια συλλογική προσφυγή με στόχο να αποστεθεροποιήσει τον ανταγωνιστή της. Προσπαθούμε εδώ να προστατεύσουμε επίσης τα δικαιώματα του καταναλωτή σε τρίτο κράτος μέλος, σε άλλο κράτος μέλος. Και για να συμβεί αυτό πιστεύω ότι χρειάζονται ενιαία κριτήρια εναρμονισμένα για όλη την Ένωση. Προτείνω κάθε καταναλωτής να δίνει την εξουσιοδότηση του να συνυπογράφει ατομικά την συλλογική προσφυγή με το σύστημα που λέγεται opt-in, Ωστόσο, εάν η αποζημίωση η οποία ζητείται τελικά είναι μικρή, ε, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να μην ζητείτε, να μην είναι απαραίτητο να έχουμε συγκεκριμένη συγκατάθεση κάθε ενός από τους καταναλωτές. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Loser Pay Principle, δηλαδή την ε, φιλοσοφία με την οποία εκείνος ο οποίος ε, χάνει την ε, δίκη θα επιβαρυνθεί και με τα δικαστικά έξοδα. Και τέλος για την προσφυγή στα δικαστήρια, για να είναι ξεκάθαρο αυτό, προσπάθησα στο κείμενό μου να ξεκαθαρίσω με βάση το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο τις αρμοδιότητες κάθε ενός δικαστηρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχουμε μπροστά μα τι συναντήσει με του σκιώδει εισηγητέ, τι οποίε θα ακούσουμε τι απόψει και τι ανησυχίε όλων. Γνωρίζω ότι η προθεσμία είναι αυστηρή για τις τροπολογίες, ωστόσο ελπίζω να αποβληθούν αυτές, έτσι ώστε να καταλήξουμε, να ψηφίσουμε το Δεκέμβριο στην Επιτροπή το κείμενο αυτό. Καταθέτω πάντως απόψε ένα κείμενο Αντιλαμβανόμενο ότι οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται, νομική, ε, ε, χρειάζονται ασφάλεια δικαίου. Ότι θα πρέπει να προστατευτούν από προσφυγέ κακή τυπίστη. πίστη. Αλλά αναγνωρίζοντα ταυτόχρονα ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα σήμερα και ότι έχουμε ενεργούς καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να προσπίσουν τα δικαιώματά του, παρεπιπτόντω όλοι οι καταναλωτέ είναι και πολίτε και ε, εκλέγουν, και οι οποίοι προσπαθούν να προστατευτούν από απαράδεκτες συμπεριφορές και καταχρήσεις της εξουσίας ορισμένων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βόλκιν έχει το λόγο. Όχι, δεν θέλετε. Η κυρία Ντελβό τότε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτη μας για την παρουσίαση της γνωμοδότησης, την οποία ανέμενα και αναμένω με ανυπομονησία. Ναι, να τη συζητήσουμε. Νομίζω ότι όλοι επιθυμούμε να βελτιώσουμε την προστασία των καταναλωτών, που το είπατε κι εσείς, είναι πολίτες που έχουν το δικαίωμα του κλαίγιν και κλαίγεστε. Οργανώσαμε ακρόαση, δεν θυμάμαι ακριβώς με πότε, την προηγούμενη εβδομάδα πάντως, και νομίζω ότι μετά από αυτό που ακούσαμε σε αυτή την ακρόαση, δόθηκαν απαντήσεις για τις διάφορες ανησυχίες, ε, ιδίω εκείνου που λένε ότι θα καταντήσουμε σε ένα σύστημα, θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα παρόνομιο με τα class actions στις ΗΠΑ. Όχι. Είχαμε πανεπιστημιακούς που μας εξήγησαν πόσο διαφορετικά είναι το, διαφορετικό είναι το σύστημα που περιγράφουμε εμεί. Υποστηρίζω την ε, εισαγωγή ε, επιπλέον έχει εγγύων ε, για τη διαφάνεια για εκείνες τις ε, οντότητες οι οποίες θα μπορούν να υποβάλουν συλλογικές προσφυγές με ένα μητρό το οποίο θα διαχειρίζεται η Επιτροπή και υποστηρίζω επίσης και την αρχή ότι εκείνος που χάνει τη, τη, δικαστική διαδικασία πληρώνει και τα δικαστικά έξοδα. Θα πρέπει Επίσης να, να, να, να δούμε τι συμβαίνει σε περιπτώσεις που ε, κάποιο ποσό δεν είχε ε, απαιτηθεί με την συλλογική προσφυγή. Σε ορισμένε περιπτώσεις έχουμε κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται εδώ και πολύ καιρό, πολύ χρόνο. Και σε ορισμένες χώρες. Και γι' αυτό το λόγο ε, όπως και εσείς είπατε, σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει έντονη κρατική επιδότηση, σε άλλα καθόλου. Γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω την πλήρη απαγόρευση χρηματοδότησης από τρίτους. Τώρα, πιστεύω ότι κατά τα άλλα το ζήτημα της, του τόπου αρμοδιότητα πρέπει να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Προέρχομαι από μικρή χώρα, χώρα. Γι' αυτό δεν είμαι σύμφωνη με αριθμητικούς περιορισμούς. 250 ίσως είναι, πολύ, ίσως είναι λίγοι, είναι μικρός αριθμός για τη Γαλλία, αλλά υπάρχουν μικρότερες χώρες στις οποίες μπορεί να είναι το σύνολο των μελών μιας καταναλωτικής ένωσης αυτός ο αριθμός. Και ε, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε τη σύμφωνη γνώμη των καταναλωτών για, το, για την εξέβρεση εξοδικαστικής συμβαστικής λύση. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας και να μην επιτρέψουμε την εξαίρεση που προβλέπεται αυτή τη στιγμή, η οποία τίνει να γίνει κανόνας. Αυτά επιγραμματικά φαντάζομαι θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όλη την προστασία των καταναλωτών στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτου δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Ε, θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι έχουμε μόνο 12 λεπτά και ένα ακόμα θέμα να συζητήσουμε. Κύριε Βόλκεν, θέλετε το λόγο? Όχι. Κύριος Ζάμετ. Σύντομος θα είμαι, Πρόεδρε. Φυσικά συγχαρητήρια στον εισηγητή για τα όσα μας παρουσίασε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό των καταναλωτών και να ε, τους ε, παρέχουμε υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όμως με τρόπο υπεύθυνο σε ό,τι αφορά ε, το ότι δεν πρέπει να ολιστήσουμε προς το αμερικανικό σύστημα. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ε, δικηγόρων που κυνηγάνε τα στενοφόρα έτσι ώστε να συμφωνήσουν ε, με τον ε, ασθενή για ποσοστά σε περίπτωση που κερδίσουν τη δίκη. Επίσης, η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται στον καταναλωτή σε αυτόν που οφείλει. Και ε, θα ολοκληρώσω με μια αναφορά στην αρχή του ε, «αυτός που χάνει πληρώνει», «χαμένος πληρώνει». Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις και είμαι σίγουρος πως τις γνωρίζει ο συγκητής που δεν είναι σαφέ ποιος κερδίζει και ποιο χάνει. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πτυχή της καλής πίστης. Ορισμένε φορές μπορεί να ε, χάσεις χωρίς, επειδή δεν μπορείς να αποδείξεις τις προθέσεις σου. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια κάποια ευελιξία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φως έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή που μας παρουσίασε την έκθεση. Ε, ως προς το περιεχόμενο, νομίζω πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Γι' αυτό πρέπει να κατεβάσουμε καλές ιδέες και γι' αυτό χρειάζεται επίσης χρόνος. Φυσικά θέλουμε προστασία των καταναλωτών και πρέπει να προσέξουμε ο καταναλωτής να βρίσκεται στο επίκεντρο και όχι όπως ε, αναφέρθηκε ε, διάφορες ε, νομικές εταιρείες οι οποίες κερδίζουν περισσότερα από αυτά που κερδίζει ο καταναλωτής. Να ασκήσω μία μικρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θέλει έτσι, επιτρέψτε μου να το πω, να ξεπετάξει τη διαδικασία. υπάρχουν περίπλοκες διαδικασίες, υπάρχει ασάφεια στο θέμα των διασυνοριακών προσφυγών και μόνο τρεις από τις 23 συστάσεις ε, που έγιναν το 2013 έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα ε, η συλλογική προστασία να μην προστατεύει τους επενδυτές αλλά τους καταναλωτές. Ήδη ο συνάδελφος ανέφερε ορισμένε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής λαμβάνει μόνο ένα κλάσμα από την αποζημίωση που δικαιούται και θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν ε, ανάγκες για σοβαρές βελτιώσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, τα κράτη-μέλη διαφέρουν ως προς τα δικαστικά του συστήματα. Στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχει ο διαμεσολαβητής, υπάρχει ο κανονισμός ε, ZPC ε, για την δημόσια χρηματοδότηση Υπάρχουν τα Ινστιτούτα των καταναλωτών, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αυτές τις διαφορές και να γίνουν διευκρινήσεις. σε γενικές γραμμές πρέπει να αποφύγουμε, να δημιουργήσουμε δυσάρεστες επιπτώσεις και να επιδεινώσουμε την θέση των καταναλωτών, να αποφύγουμε την ε, αναζήτηση ευνοϊκής δικαιοδοσίας και να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια για τις εγκεκριμένες οντότητες. Το άρθρο 4. Επίσης, ε, να υπάρχει δυνατότητα opt-in, άρθρο 6, για διασυνοριακές προσφυγές και εμπορικές, ε, και εμπορικές επενδύσεις, άρθρο 7. Και εκεί χρειάζεται προσοχή. Επίσης, οι απολαβές των δικηγόρων θα πρέπει να ε, διευκρινιστούν έτσι ώστε το πρώτο μέλημά μας να είναι προστασία του καταναλωτή και όχι το κέρδος των ε, νομικών εταιρείων. Αυτά έτσι εν συντομία. Θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερες παρατηρήσεις, αλλά θα περιοριστώ στο να αναφερθώ σε αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόλκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θέλω να πω κάτι εν τέλει. Ήμουν σε μία άλλη ακρόαση πιο πριν Και στις 10 Οκτωβρίου λοιπόν, οι καλεσμένοι ήταν έξι νομίζω, είπαν ότι ε, πρέπει να προσέξουμε και να αποφύγουμε, να καταλήξουμε, ε, να γίνουμε μερικοί με τη συλλογή, στο θέμα των συλλογικών προσφυγών. Ε, και εγώ έχω πολλά να σχολιάσω, όμως ε, να πω καταρχάς ότι αυτή η πρόταση της Επιτροπής δεν θα μας οδηγήσει σε μια βιομηχανία προσφυγών όπως γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε και πρέπει να ε, αποβάλουμε αυτήν την ε, ιδέα, γιατί αυτά είναι μύθος, δεν είναι αλήθεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικό οι περισσότερες πολιτικές ομάδες να τοποθετηθούν. Δεν είμαστε εδώ να προωθήσουμε παραγωγική διευθέτηση διαφορών ή καταχρηστική όπως οι Αμερικανοί. Δεν το θέλει κανείς αυτό. Δεν είναι ο στόχος μας. Τι μπορούμε να δούμε. Όσον αφορά τους ε, εγκεκριμένου φορείς, όπως είπε και ο εισηγητής, πρέπει να εντάσσονται σε μια διαφανή διαδικασία. θα πρέπει και κάποιοι φορείς να διαμορφώνονται ad hoc κατά περίπτωση. Δεν θα περιοριζόμουν μόνο σαν ανεξάρτητους δημόσιους φορείς και προσώπους ε, καταναλωτών. Σε κάποιες ακροάσεις ακούσαμε καλές εθνικές πρακτικές και ο κύριος Φως αναφέρθηκε στο συνήγορο του πολίτου στη Δανία και τη Φιλανδία. Εκεί λειτουργεί εύρυθμα το σύστημα, μπορούμε να το δούμε. και την αρχή που πληρώνει αυτός που χάνει. Την αμφισβητώ για τους λόγους που ανέφερε και ο Ζαμίτ για το πεδίο εφαρμογή. Συμφωνώ με τη Μαντίν Τελβό. Μπορούμε να το διευρύνουμε το πεδίο. Έχω υπόψη μου κάποιες εθνικές πρακτικές που καλύπτουν τα θέματα διάκρισης και ισότητας, κυρίως στο χώρο εργασίας. Άλλος τομέας είναι οι περιβαλλοντικές βλάβες θα πρέπει με σοβαρότητα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο διευρύνσεως του πεδίου εφαρμογή. Ευχαριστώ. Λόγω χρονικών περιορισμών περατούτε η συζήτηση του σημείου 13. Πάμε στο σημείο 14. Oh, sorry, my, my, my mistake. Uh, deadline... Λάθος, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 5 Νοεμβρίου. 5 Νοεμβρίου. Μην ανοίξουμε κουβέντα τώρα. Όχι. Όχι. Do, do agree on Συμφωνούμε με τις 7, 7 του μηνός. Κύριε Γκυγγί, είμαι υπέρ να μπορούμε να καταθέσουμε μέχρι 7 Νοεμβρίου, αν δεν υπονομεύσουμε όμως το χρονοδιάγραμμα που προανέφερα. Στόχο ψηφορία στην Επιτροπή το Δεκέμβριο. Συμφωνώ. Αλλά θέλαμε να σίγουρος ότι δεν θα αναβληθούν τα υπόλοιπα στο χρονοδιάγραμμα. Δεν νομίζω με δύο μέρες γίνεται ζημιά. Συμβιβασμός. Να πούμε στις έξι. Μου λέει η γραμματεία ότι διαφορετικά θα υπήρχαν προβλήματα. Έξι. Ωραία. Έξι. Σημείο 14. Πρωτόκολλο 3. Ο κ. Σπέλκαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα πω πολύ γρήγορα και ελπίζω να μην ε, είναι αυτό πρόβλημα για τους διερμηνείς. Έχει να κάνει με την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος είναι καλύτερη ένωμη προστασία στην Ένωση. Νομίζω πως όλοι έχουμε αυτόν τον στόχο. Η πρόταση λοιπόν του Δικαστηρίου είναι, πιστεύω, μία πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται μία τροποποίηση σε θέματα ορολογίας της συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό το θεωρώ πολύ συνετό. Ως προς το περιεχόμενο τώρα, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις ε, προσφυγικών ακύρωσης είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 262 ή 3 της ε, συνθήκης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ε, κυρώσεις και τα πρόστιμα. Μετά αναφέρονται οι περιπτώσεις ε, της διαδικασίας σε παραβάση και οι προσφυγές ακυρώσεως που θέλουν να μεταβιβαστούν στο Γενικό δικαστήριο. Ε, δεύτερο σημαντικό σημείο αφορά τη δημιουργία μίας διαδικασίας έγκρισης η οποία αφορά περιπτώσεις ε, τις οποίες ε, οι οποίες χρήζουν ε, εξέτασης, επανεξέτασης. Εδώ προτείνεται η δημιουργία μίας ανεξάρτητης αρχής. Χρειάζεται η συνεισφορά και σύμφωνη των κρατών μελών διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νομικό ζήτημα για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ ε, δεν αναφέρεται αυτή η αρχή, υπάρχει μόνο μία γενική αναφορά, υπάρχει κάποια ασάφεια, χρειάζεται λοιπόν διευκρίνηση και νομίζω πως ε, πρέπει στο κείμενο να αναφέρεται ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου, είτε αυτές είναι ε, θετικές τα αρνητικές πρέπει να συνοδεύονται από κάποια αιτιολόγηση. Το δικαστήριο στο, στην πρόταση του έχει επεξεργαστεί την ε, αρχική του πρόταση και η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ε, αφορά την ε, θέση ισχύ τον Δεκέμβριο του 2020 της νέας ε, μορφής λειτουργίας του. Θεωρώ πως και αυτό είναι εύλογο και σκόπιμο για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Ε, αναφέρεται η αύξηση του αριθμού των δικαστών. Ε, επίσης, χρειάζεται να αναφερθεί πως ε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και στην ίση ist. Das ist praktisch, aber die Kommission wird sicherlich ähm, schriftlich beantworten können. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα τα οποία έχουν ε, μείνει αναπάντητα από την Επιτροπή. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας τα απαντήσει και τέλος ερώτηση στην Επιτροπή πότε σκοπεύει να δημοσιεύσει την δική της πρόταση γιατί κύριο μέλημά μας είναι οι πολίτες της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φως. Και εγώ θα είμαι σύντομο. Εκ μέρου του κυρίου Ράντεφ, ο οποίο είναι σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πρότασή του, για το σχέδιο έκθεση. Η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου είναι κάτι το αναγκαίο και ο κύριο Ράντεφ υποστηρίζει επίση την θέση του κυρίου Βόλκεν για την ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων στην σύνθεση του δικαστηρίου. Δεν πιστεύει όμως ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, έτσι όπως το προτείνει το δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσει τις δικές του τροπολογίες. Επίσης, ε, συγχαίρει τον κύριο Βόλκεν και τους υπόλοιπους κοιότητες για την άριστη συνεργασία. Και ευχαριστεί για ε, τη συνεργασία. Άλλη μια φορά. Δεν έχουμε εκπρόσωπο του δικαστηρίου. I guess, ε, so the deadline for... Προθεσμία υποβολής τροπολογιών. 31 Οκτωβρίου του 2018 στις 5 το απόγευμα. Για το σημείο 14. Ευχαριστώ. επόμενη συνεδρίαση. Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου. Και ευχαριστώ τη διερμηνή που μα έδωσαν και άλλο χρόνο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα. Γεια.